κείμενο. Ωραία. Θα το καταγράψουμε. Άλλο διαδικαστικό. Παρακαλώ. Το ίδιο πράγμα και εγώ, Πρόεδρο. Στη Ρωσία υποστήριξε το ψήφισμα, αλλά δεν ε, χτύπησε το μηχάνημα. Ευχαριστώ.